Good evening, ladies. Is One, two. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλετε να περάσετε ώρα στο Στρασβούργο ή να πάτε γρήγορα στα δωμάτια του ξενοδοχείου σας. Λυπούμε που οργάνωσα σήμερα, απόγευμα Δευτέρα Στρασβούργου, αυτή τη συνεδρίαση. Δεν είναι η πιο βολική ώρα, έχουμε όμως πάρα πολλές ψηφοφορίες που πρέπει να διεκπαιρεώσουμε. Θα προσπαθήσω αυτό όμως να μείνει εξαίρεση και να μην γίνει κανόνας, δηλαδή συνεδριάσεις Δευτέρας. Έγκριση μερσιας διάταξη. Έχετε σχόλια, όχι. Επομένως, εγκρίνεται η μερισία διάταξη. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου δεν έχω κάποια ανακοίνωση, οπότε μπορούμε να περάσουμε ήδη στο σημείο 3, την πρώτη ψηφοφορία, σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Πρέπει να πω ότι η έκθεση για την γνωμοδότηση αυτή είναι εξαιρετική. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, έκανε πολύ καλή δουλειά. Δεν θέλει να πει ο ε, κάτι περισσότερο. Εσείς, αν όχι, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Okay. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λιτολική αναφορά 1. Citation 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Περνάμε στην 85 τροπολογία. Απορρί... Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Α, δεν το είπα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, το ξαναλέω. Τη αναφορά 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 85 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 86. Άρχεται ψηφοφορία. Machst hier an? working? 49 είναι παρόντες, έχουν ψηφίσει 48 εξ αυτών. Πέρας. Εγκρίνεται η 86. 106 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 ψήφι πέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν τέσσερα ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Όχι. 108 ψήφι περ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 114 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 115 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 117 μου λένε ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 10 ψήφι υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε τη 10 Άρχεται ψηφοφορία. Δεν θέλω να, είμαι, να επηρεαστώ. Λοιπόν, γι' αυτό ζήτησα έλεγχο. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά αποχές, Ελέγχουμε την 120. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 121 ψήφι περ. κατά αποχές εγκρίνεται 122 ψήφι περ. κατά αποχές απορρίπτεται 123 ψήφι περ. κατά αποχές απορρίπτεται 124 ψήφι περ. κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 124 Καστάλτο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σαφές απορρίφθηκε. 125 ψήφι περ, κατά αποχές απορρίπτεται. 126 λόπες περ, κατά αποχές. 129 ήταν, ναι. Εντάξει, εντάξει. 128 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 128 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Μα σαφώς απορριπτόταν. Απορρίφθηκε λοιπόν. 130 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν είμαστε σίγουροι, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 126. Πέρας. Εγκρίθηκε. Σαφώς. 127 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 127 του κύριου Πάσκου. Πέρας. Απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά αποχές, τι κρίμα, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 135-136 ψήφι υπέρ, κατά Αποχές. Απορρίπτονται. 137 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 138 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 139 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 140 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται ευτυχώς. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, εποχές, Εγκρίνεται. 173 Βαλέρο. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 175 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 174 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177 ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 178 ψήφι πέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 179 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 180 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε την 182, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 183 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 184 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 185 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην 187 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται.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 Τέλο πάντων, είχε καταπέσει. Ναι, είχε καταπέσει. 201 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Έτσι πρέπει τουλάχιστον αλλά ας ελέγξουμε τη 205, άρχεται η ψηφοφορία. 205, Λίτς Κρέλ Φρόιντ. και άλλοι. Απορρίπτεται σαφώς. 206 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 207 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 208 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 209 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 212 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 215 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στη 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τι ωραία. 218 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 220 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε τη 220 άρχεται η ψηφοφορία It's closed. This Πέρας απορρίφθηκε. 221 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 224 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 225 υπέρ, κατά αποχές. Θα ελέγξουμε το 225, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 226 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 231 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 230 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 232 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 233 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.34 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε τη 2.34, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 26 υπέρ, 25 κατά. Αυτά. 2.35 υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται. 2.36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.38 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.39 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 2.41 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.42 υπέρ, κατά αποχές, θα ελέγξουμε τη 2.42, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε ξεκάθαρα. 2.43 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 2.44 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.45 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.46 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.47 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.48 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 2.49 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τι έγινε με την 106, έχει αποσυρθεί, έχει απορριφθεί, άρα δεν ψηφίζουν. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τη 253 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 2.54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.61. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και πού πηγαίνουμε τώρα. Στην 21, πολύ ωραία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 καταπίπτει και πηγαίνουμε στην 26. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε το 29 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 32 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καστάλθο, 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εκρίθηκε. 37. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 42 και 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 44 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται.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 Εγκρίνεται ωραία και αυτή. 63. Η Φανόρντιν. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 67. 27. Μάλιστα. Έχει εγκριθεί 106 Μάλιστα. Εντάξει, κατάλαβα. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξω την 75 άρχεται ψηφοφορία Closed. This has been clearly rejected. Πέρασε. Ψήφο απορρίφθηκε. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά απόχέ, απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά απόχέ. απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά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 Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το 4, στρατιωτική κινητικότητα, εισηγητής του Νεκέλαμ. Θα θέλετε να πάρετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές ε, για την επικοδομητική και θετική συνεργασία. στόχος αυτή της έκθεσης είναι το να δώσει έντονα πολιτικά κίνητρα για τις χώρες μέλη προκειμένου να επιταχύνουν την αμοιβαία συνεργασία, να υπάρχει ετοιμότητα προκειμένου να επιτευχθεί η στρατηγική κινητικότητα. Γιατί η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο και θα έχουν πρακτική, όλα αυτά πρακτική αξία. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας και για την ε, βούληση που επιδείξατε να το στηρίξετε. Ευχαριστώ τον Νίκ Κέλαμα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα αίτημα από την σοσιαλιστική ομάδα. Μου ζητήθηκε να υποβάλω μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία 6 προκειμένου να αντικατασταθεί το end introduced reinforcements from outside με το συμπεριλαμβάνοντας τις εξωτερικές συμμαχικές δυνάμεις, including external allied forces. Ε, δεν μπορώ να δεχτώ την τροπολογία. Θα μπορούσα να δεχτώ την τροπολογία εάν δεν υπάρχει αντίρρηση από τέσσερις συναδέλφους. Αντιρρήσεις όχι μπορούμε να τη δεχτούμε συνεπώς. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συμβαστική πρόταση 10. Υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται. 77. Υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται. 78. Υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται. 80. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 11. Υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται, 89 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται. Η 90 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ, κα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 ε, ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ εγκρίνεται. 190-120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική η πρόταση 20 υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 146 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 146 αρχή της ψηφοφορίας Απορρίφθηκε. 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152. Υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε την 153 Αγιάλα σέντερ Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας σαφώς έχει απορριφθεί. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν ψηφίζουμε την 155-156 ψήφι υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 156 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 171. Ψηφίζουμε. υπέ, ε, ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Εκτιμώντα, υπέρ, 4 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 5 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 6. Ως, όπως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 13. κύριο Νταζάν υπερκατάποχη. 30 ε, για, για, να ελέγξουμε την τροπολογία 30. κύριο Νταζάν αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 αποσύρθηκε τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 47 κύριος Νταζάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 ε, ε, συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται 7 ε, ε, υπέρ κατά 8 εγκρίνεται. Περνάμε στο 56, κύριο Τανόδου, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, υπέρ κατά αποχές. Για να ελέγξουμε το 58. 58. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 59 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμπεριστική 9 υπέρ κατά ε, ε, εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 67. Ψηφίζουμε για την 67. Απορρίφθηκε. 67. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης ε, είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία λοιπόν της έκθεσης, αρχίζει η ψηφοφορία. Μπορούμε να τελειώσουμε, ε, να την ε, κλείσουμε 39 υπέρ 13 κατά. Παρακαλώ. Θα Θέλαμε να υποβάλουμε μια έκθεση μειοψηφία και την έχουμε ήδη υποβάλει στη γραμματεία. Ωραία, ευχαριστώ. Περνάμε στο 5, ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Ο κύριος Πάσκου, παρακαλώ, θα θέλετε να πάρετε το λόγο και μετά να ψηφίσουμε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 26. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτηκε. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά για να ελέγξουμε την 37 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ για να ελέγξουμε τη 38 για να ελέγξουμε τη 38 Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Σαράντα υπέρ κατά αποχές Ναι, για να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμπατησχίδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε, 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε, 55 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε, 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τη τρολογία του Κεφαλογιάννη, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 58 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε με την 8. Υπάρχουν δύο συνάδελφοι. Πέρας ψηφοφορία εγκρίθηκε. 59 υπέρ, κα, κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 72 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 72 αρχίζει η ψηφοφορία απορρίφθηκε Εξεπτά, αν υπέρ κατά εποχές ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχή πέρας πληροφορίας απορρίφθηκε. Ε, 66 ρογεύση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, να ελέγξουμε. Για να ελέγξουμε την 66, Τροβεύσκη. Πέρας φορείας. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Περνάμε στην Κλέρ Μούντι. 68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75-76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70, 80 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά Ποχές απορρίπτει, 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει, 74 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 84. 84. η κ. πέρας απορρίφθηκε. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91. Μαμίκες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 την αποσύρεται. 158 ζώνιες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αποσύρεται του κυρίου Πάσκου, 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την 112 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, 25 κατά, 18 κατά, υπέρ, ε, 25 ε, υπέρ κατά, ποιες εγκρίνεται. Δεν υπέρ κατά, 121, 22, υπέρ κατά, ποχές εγκρίνεται. 122. Θα έλεγα, θα, έλεγα, θα έλεγα ότι εγκρίνεται, εν πάση περιπτώσει, ξαναψηφίζουμε. 122. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όχι. 123. Να ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Σαφώς απορρίφθηκε. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 128 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 128, αρχίζει η ψηφοφορία. πέρα ψηφοφορία. εγκρίθηκε. καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει. Έχουμε φτάσει στην 133. 133. Ράντος, άλλοι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές και απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140-141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 148 Τώρα ε, ε, ε, υπέρ κατά αποχές σαφώς εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές 143 για να το ελέγξουμε αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την 149 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίθηκε. Αύκο 8 υπέρ κατά Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156. Μίκης, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 166 του κυρίου Νταζάν η δεύτερη ευκαιρία πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε και πάλι Βασική ψηφοφορία 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε επιτέλους. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τη 276 θα πρέπει να την ψηφίσουμε ξεχωριστά. Πάμε Πρώτα στην 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αύκο 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία του 176. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε την 176. Ναι ή όχι. Πέρας πληροφορία Σαφώς απορρίφθηκε. Συμβαστική 11. Υπέρ κατά ε, ποιες εγκρίνεται 100, ε, ε, υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 185 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 184 κατά πίπτη 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189, 190, 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 για να ελέγξουμε, 208, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε τη 215 ψήφι υπέρ. 2, 2.16 υπέρ. Κατά ποχέ εγκρίνεται. 2.17 υπέρ. Κατά ποχέ απορρίπτεται. 2.18 υπέρ. Κατά ποχέ εγκρίνεται. 2.19 υπέρ. Κατά ποχέ εγκρίνεται. 2.20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά ποχέ εγκρίνεται. 2.26 κατά, υπέρ κατά για να ελέγξουμε τη 226 αρχίζει η ψηφοφορία 226 Λείπουν λοιπόν, δύο συνάδελφοι πέρας ψηφοφορίας. 27, 27. 27 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Πού είμαστε τώρα? 2.56. Τροπολογία Πάσκο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται κύριε Πάσκο. 2.27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.42 υπέρ κατά αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Να έρθει ο Έλμερ. Πέντε συνάδελφοι απουσιάζουν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 2.43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.45 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2,47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, θα το ε, επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 2.57. Πέρασα. Ε, εγκρίνεται με μικρή πλειοψηφία. 2,59 καταπίπτει. 2,63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2,61 ήταν η προηγούμενη. 2,62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2,64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2,65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αύκο 9. Υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς. Ψηφίζουμε την 9 της Επιτροπής Θεματικών Υποθέσεων. Αύκο 9. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική. Η 258 εγκρίθηκε. Καλώς. Καταρχάς, ψηφίζουμε την 9 της ΑΦΚΟ, αυτό απορρίφθηκε. Τώρα με ενημερώνουν ότι κάναμε ένα λάθος και πρέπει να ψηφίσουμε τη 259. Κύριε Πάσκου, σας αφορά. Σας ζητώ συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ του κυρίου Πάσκου και της τροπολογίας του 259. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 259. Πάμε τώρα και επιστρέφουμε στις μυστηριώδεις ε, ψηφοφορίες των τροπολογιών της ΑΦΚΟ. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 της ΑΦΚΟ. Υπερκατά αποχές εγκρίνεται. 7 της ΑΦΚΟ. Υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 10 της ΑΦΚΟ. Υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώ τη 10 τροπολογία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων τη ΑΦΚΟ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τρει συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές αναφορές. Η ένα, Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η δεύτερη εγκρίνεται. Η τρία Υπέρ κατά εγκρίνεται, η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Κυρία Λέζιν για θέμα διαδικαστικό, παρακαλώ. Η ομάδα μου θέλει να υποβάλει έκθεση μειοψηφία και προφορικός να τη διαβιβάσει στην γραμματεία. Και σας ευχηστώ την προσοχή στο γεγονός τούτο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Λόισεν. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 6 ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα σχετικά. Η εισηγητής είναι ο φίλος κύριος Πέτρας Αουστρεβίτσιους. Θέλετε το λόγο παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους κοιόδης εισηγητές για την πραγματικά εξαιρετική τους συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και τους εμπειρογνώμονες και τους ειδικούς που συμβουλευτήκαμε για την πολύ αποτελεσματική στήριξή του, στήριξη όλων αυτών των ε, στελεχών. Νομίζω ότι η έκθεση αξίζει την υποστήριξη όλων και γι' αυτό σας καλώ να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Ας μπούμε στο ψαχνό λοιπόν. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται η συμβαστική 2. Πάμε στην 2 τη επιτροπή Γενικών. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φάμε 27. υπέρκατα κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. υπέρκατα, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. υπέρκατα, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. υπέρκατα, κατά αποχές εγκρίνεται. Φανταστική έκθεση. Συμβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120. Κύριε Πώς, δικιά σας τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Να το δούμε ηλεκτρονικά. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 120 τροπολογία του κύριου Πώς. Πέρασε. Εγκρίνεται σαφέστατα. 121 και 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ, υπέρ, όχι, όχι, κρίμα, πολύ κρίμα. Λοιπόν, Ελπίζω να σας πιάσω στον ύπνο. Την 145 του κύριου Κοράου, να την ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 155, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε... Α, να την ελέγξουμε την 155, της κυρίας Βεργιά. Ψηφίζουμε την 155 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία 157. Πέρας. Εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφοφορία κατά τμήματα στη 206. Το ζήτησε το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 206. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της Ετροπολογίας 206. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται και αυτό. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 219 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν Δεν έχουμε τροπολογήσει από την Επιτροπή ΦΑΜΑ, γυναικών. Καλό, συμβαστική 24. Υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την συμβιβαστική τροπολογία 24. Πώς ψηφίζουμε. The vote Now closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Σαφέστατα εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην ε, τέσσερα τροπολογία της Επιτροπής ΦΑΜ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 της ΦΑΜ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 278 τροπολογία του κυρίου Μικολάσικ. Υπέρ κατά αποχές. Θα το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 278. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 334. Α, καλώς. Συμβιβαστική 32, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα στην 334 με την προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασα. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 εννοεί ο πρόεδρος μάλλον. Τη 34. Ψηφίζουμε τώρα την 346 ε, του κυρίου Βάγκελ. Υπέρ, ε, εγκρίθηκε. 352 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 35 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική 35. Πέρασε. Σαφέστατα εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα στην 377. Γιατί αποσύρθηκαν οι προηγούμενες. Κατανοώ. Ποιος είναι υπέρ τη 377. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 382 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβιβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στη συμβιβαστική 43. Καλώς. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, τροπολογία μάλλον 52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία υπαριθμών 1. Πέρας. Εγκρίθηκε. Καμία ψηφοφορία για τη 2. Ψηφίζουμε την 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ κατά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 θα την ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 15 του κυρίου Βάγκελ. Πέρασε. Εγκρίνεται σαφέστατα. 16 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία της κυρίας Βερσιά. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 20. Πέρασα. Εγκρίθηκε. 21 καταπίπτει. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 25. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 31 και 32 καταπίπτουν. Πάμε στη 33 της κυρίας βεχσιά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 33 της κυρίας Βεχσιά. 33 ή 32. Την 33, πολύ σωστά. Την 33 ψηφίζουμε. Πέρασε ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εγκρίνεται η 33. Δεν εγκρίθηκε η 4, άρα ψηφίζουμε την 34 της κυρίας Βεωσιά. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 35, υπέρ, κατά, αποχές. Το ελέγχουμε. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 36. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Η 35 εγκρίθηκε, γι' αυτό και πάμε στην 38. Της κυρίας βεχσιά και πάλι. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 39 ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Με ενημερώνουν ότι πρέπει να πάμε στην τροπολογία 34 που έχασα της κυρίας Βερσιά. Ψηφίζουμε την 34 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 30 εγκρίθηκε. Πάμε στη 41. Υπέρ κατάποχες εγκρίνεται. Η τελευταία καταπίπτει και γι' αυτό ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 41 ε, υπέρ 6 ψήφοι κατά. Έχω λοιπόν τώρα κάποια θλιβερά νέα για σας. Ε, φτάνουμε στην τελευταία ψηφοφορία. Κάτι που σας στενοχωρεί πολύ. Το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Σχέδιο έκθεσης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία. Ο ε, Μάικλ Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Χαίρομαι γιατί βρήκαμε ευρείες συμβιβαστικέ ε, λύσεις ε, για όλες τις τροπολογίες. Έχουμε περιορισμένο κείμενο, πολλά θέματα θα μπορούσαμε να τα έχουμε συμπεριλάβει γιατί έτυχαν ευρεία συνένεση κατά τη διάρκεια τη σύνταξη τη έκθεση αυτή και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερω διότι το πράξαμε και προσπάθησα να συμπεριλάβω και θέσει συναδέλφων που τελικά δεν θα μπορέσουν να την υπερψηφίσουν την έκθεση αυτή. Ωστόσο, εάν κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν, για παράδειγμα για τον τομέα των ε, κοινωνικών υποθέσεων και των εργασιακών, τότε θα πρέπει να αποτελούν μέρο τη έκθεση αυτή. Προσπάθησα δηλαδή να είμαι θετικό, να συμπεριλάβω όλε τι απόψει και βεβαίω είμαι ανοιχτό σε οποιαδήποτε κριτική, επίκριση ή σχολιασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Μάικλ Γκάλερ. Αν δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο, ξεκινάμε.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 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73 έχει αποσυρθεί. 74 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 από τον Τσίτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 πάει υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά εποχέ. απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε 114 πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14, Λέω. Συγγνώμη, 13, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 14, συμβαστική υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 120 σαφοζέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ, Κατά. Έχει αποσυρθεί 121. Δεν το έχω στο κατάλογο. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 122 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 128 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 129 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Favor. Against. κατά εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 164 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε την 165 έκτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 166 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69 was adopted, so 167 για την κρίση 69. 169 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 173 και 174 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Στις ε, υποκατηγορίες 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το και 1α υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Προφορική ένα αλφα Κατά αποχέ εγκρίνεται. 10 αποχές Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική ένα υπερ κατα αποχές εγκρινεται δέκα υπερ κατα αποχές εγκρινεται συμβαστικη ένα υπερ κατα αποχές εγκρινεται συμβαστικη δύο υπέρ. αποχές αποχέ εγκρίνεται. δύο 2α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Οχ. Of course. Μα βέβαια, πώς ξέχασα. Πίτσουλα, 28 υπέρ, κατά, εποχές. Θα ελέγξουμε κιόλας την 28. Πέρα συγκρίθηκε. 29. Χαβιέρ Νάρτι, πέρ. Κατά. Οποχές. Θα φτελέξουμε και την 29. Πέρας. Απορρίφθηκε. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται συμβαστική. Να ελέγξουμε. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική 2. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Γκάλερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 38. Ε, ας το ελέγξουμε τέλος πάντων. It's Πέρας. Απορρίφθηκε. Τολογικές αναφορές. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ίντα. 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ίντα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα τρία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα τέσσερα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και φτάνουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία του συνόλου του σχεδίου όπως έχει τροποποιηθεί. Καλά είπα. Ναι, άρχεται η ψηφοφορία. And it is closed. Πέρασε. Εγκρίθηκε 41 ψήφοι πέρα, 9 κατά και μία αποχή. 9. Επόμενη συνεδρίαση. ένα είπα, 9. Λοιπόν, επόμενη συνεδρίαση, 21 και 22 Νοεμβρίου. Δεν πιστεύω τολμάει κανείς να πει ε, τίποτα για τα διάφορα. Όχι. Επομένως, 8.30 ακριβώς και λήξαμε.